Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΠΑΜ και και όλους τους αναπληρωτές. Παρακαλώ καθίστε. Καλημέρα στην ε, πολυάριθμη επιτροπή μας. Έχουμε κοινή συνεδρίαση ΦΑΜ και ΝΤΕΒΕ σήμερα το πρωί. Και έχουμε μια μεγάλη, ένα μεγάλο κατάλογο ψηφοφοριών. Να ευχηθώ ένθερμη καλημέρα στον κύριο Τομπέ. Και έχουμε την ε, τιμή να συμπροεδρεύσουμε για μια ακόμη φορά εν ώψη αυτής της νέας ε, νομοθετικής περίοδου θα έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι. So sorry to push now a little bit, but we, we have a long list uh, and I know... Με συγχωρείτε που σας πιέζω, έχουμε μακρύ κατάλογο και ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος ε, και τους συναδέλφους. Καλωσορίζω λοιπόν τα μέλη της ΦΑΜ και της ΔΕΒΕ. Καλημέρα σας ε, και καλή χρονιά σε όσους δεν έχω συναντήσει ακόμη. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας και είναι πολύ καλό σημείο αφετηρίας ε, Ας ε, περάσουμε και στις ψηφοφορίες και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέγνερ γιατί έχουμε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών μας. Τα βλέπετε και στα αποτελέσματα και ελπίζω να δώσουμε και ένα ισχυρό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με τα λόγια αυτά, ας περάσουμε στην ημερησία διάταξη και θα περάσω στα γερμανικά. Παρακαλώ, φορέστε τα ακουστικά σα. Έγκριση τη ημερήσια ε, διάταξη. όσο δεν χρειάζεται κάποια αλλαγή να γίνει. Also, <laughs> also wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Να περάσουμε στο 2 της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, αν δεν υπάρχουν ε, αλλαγές, θεωρείται εγκεκριμένη η ημερήσια διάταξη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ένταση. Ελπίζω να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα τώρα. Μάλιστα. Ακούω ότι δεν χρειάζεται να σας ε, ανακοινώσω τις ανακοινώσεις της Προέδρου, γιατί τα διαβάζουν και τα μέλη τη Επιτροπή ΔΕΒ. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Και άρα γλιτώνουμε χρόνο. Και έτσι λοιπόν μετά τι ψηφοφορίε θα κάνουν τι ανακοινώσει στα μέλη τη Επιτροπή ε, ΦΑΜ. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να περάσουμε παρά αυτά στι ε, ψηφοφορίε. Μαζί με την ε, Επιτροπή ΜΑΝΤΕΒΕ, η 25η επέτειο τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη στο διάσκεψη του Νερόμπι. Ε, καταρχάς σχέδιο προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε λοιπόν. Η τελική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν ε, ε, είμαστε σίγουροι για αυτό το αποτέλεσμα. Παράγραφος 1. Παράγραφος 1 ψηφοφορία κατά τμήματα, την οποία την έχει ζητήσει η ομάδα του ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα. Όλη η παράγραφος χωρίς Sexual and Reproductive Health and Rights. Η κοινή αποστολή λοιπόν για τους Έχετε όλα τα στοιχεία μπροστά σας. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Και εδώ ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα από το ΕΛΚ. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγράφος 5 πάρει ψηφοφορία κατά θνηματά, Πάλι ζητήθηκε από την ομάδα του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν έτσι στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Μία ψήφος υπολείπεται. Αν ψήφισατε όλοι σας λοιπόν τώρα. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίνεται. Σχέδιο προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι στην παράγραφο 1, παράγραφος 1, μετά από έτοιμα ε, της ε, του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. 4. Και πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της παραγράφου 4. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και εδώ, για την τελευταία τελική ψηφοφορία, θα κάνουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία. Έναρξη παρακαλώ. Πέρασε. Και πάλι με συντροπτική πλειοψηφία εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στο σχέδιο α, ψηφίσματος. Παράγραφος 1. Η 88 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 9. Για την παράγραφο 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Συμβαστική 10 τώρα. Υπέρ. Η συμβαστική 10 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην 101. προπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 127. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 106. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται η 108 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται Παραγράφος 4 σε τμήματα ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ υπέρ κατά άποχες Εγκρίνεται. 109. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Να περιμένουμε λίγο ακόμα. Τώρα ψηφίσατε όλοι σας. Πέρα ψηφοφορίας λοιπόν. Έγκρινεται. Και περνάμε τώρα στην 110. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 111. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112, 113 και 114. Ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Μας λείπει ακόμα μία ψήφος. Πέρα ψηφοφορίας. 20 είναι υπέρ, 16 κατά εγκρίνεται. Για 118 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Μάλλον είμαστε πλειοψηφία, αλλά να το ελέγξουμε παρακαλώ. Την 118 παρακαλώ, την ε, επιβεβαίωνουμε, την επαληθεύουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Καταπίπτει. Η επόμενη. Απορρίπτεται και αυτή. Απορρίφθηκε, συγγνώμη. Άρα, η 132. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 133. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 135 και 138 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 137. Έναξη ψηφοφορίας. 23 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, εκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην παράγραφο 9. Α, συγγνώμη. Έχουμε πάει παρακάτω. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139. Υπέρ. Α Ας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά γιατί δεν είμαι σίγουρη. Την 139 παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη. Πέρας. 34 κατά, 9 κατά. Ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, αλλά δεν είδα τα χέρια σας παρακαλώ, έτσι πως τα σηκώνονται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 142. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στη συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 192. Υπέρ. Κατά. 192, ναι. Στη σελίδα 9. Υπέρ. 192. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 και 170 που είναι ταυτόσημες. υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15. Κάποιες σελίδες παραπέρα στη σελίδα 13. Υπέρ. Για τον συμβιβασμό υπερασμό 13. 15, συγγνώμη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 18. Παράγραφος 18 με χωριστή ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚΑ. Υπέρ. Παράγραφος 18. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 185. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186. Υπέρ. Κατά. Ναι, συγγνώμη. Η 186. Άλλη μια φορά. Παρακαλώ να δοκιμάσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 172, 189, 190. Από κοινού, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 και 194 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κατάλογος ψηφοφορίας έχει πολύ ακόμα. Ναι, θέλω να σας... Είστε υπομονωτικοί. 197. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 198. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 200. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Η 201. Α, συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Η 202 παρακαλώ, λέει η πρόεδρος. Όχι. Εγκρίνεται. Η 202 παρακαλώ υπέρ για τη 202 κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 16 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 167 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Recitals. 16. Αιτιολογική σκέψη α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 με σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Για την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 και 22 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και έτσι περνάμε στην 27. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται στην τριάδα να περάσουμε λοιπόν τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 στις απ' σκέψεις πάντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Ε, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τριάντα οκτώ. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία τρίαντα 38 στην αιτηλογική σκέψη F. A. Μας λείπει μία ψήφος. 15 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. Και να περάσουμε στην συμβαστική 3, ε, λογική σκέψη G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι, δεν θα ψηφίσουμε το 49, αλλά πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Εντελογική σκέψη IA. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη είναι η τροπολογία 65. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη π. Ρόλινγκο. Καταπίπτει. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος. Και φτάνουμε στην ετυλογική σκέψη R. 77 Τροπολογία 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78. Ο κ. Τραμπέλα, κάτι διαδικαστικό. Για ποιο λόγο ε, καταπίπτει συνέχεια, καθώς ε, ε, έχει απορριφθεί η 76, γιατί λέει καταπίπτει ε, αν υιοθετηθεί η 76, ενώ απορρίφθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε για τα δύο μέρη του κειμένου, κατά την απόψή μου. Ναι, και εγώ αυτό έλεγα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα κύριε Τραμπέλα. Να ψηφίσουμε λοιπόν την αθλητική σκέψη π. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Wir zu 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στο S79. Τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΤΑΦ 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιου, Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται, διορθώνει η πρόεδρος. Εγκρίνεται. Και έτσι περνάμε στην 85, τροπολογία 85, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 86, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται τώρα περνάμε στα citation. Ένα τροπολογία 1. Υπέρ. Βλέπω ότι είναι ταυτόσιμη με τη 2. τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Να ελέγξουμε. Έναρξη. Παρακαλώ, ηλεκτρονικά την τροπολογία 3 στις εκλογικές αναφορές. Πέρα ψηφορίας. 25 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στη συμβαστική 1, στις λειτουργικές αναφορές, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7. 12 και 13. είμαι. Υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Με τα χέρια σα. Υπέρ παρακαλώ τροπολογία 8. Ε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 10. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Έγκρινεται. Η 14. Α, συγγνώμη, λέει πρόεδρο, συγγνώμη. Εγκρίθηκε η συμβαστική υπαριθμών 2 και έτσι μετά από μια μακρά ψηφοφορία να περάσουμε και στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Yeah, yeah, Πέρας ψηφοφορίας. Και όπως βλέπετε, 39 είναι οι ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά, 3 οι αποχές. Να, μας συγχαρούμε, να σας συγχαρώ όλους σας, να σας συγχαρώ για την ενεργή συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, ψηφοφορία. Και να ευχαριστήσω και τους συναδελφούς της Επιτροπής Ανάπτυξης για τη συμμετοχή τους. Και θα ήθελα και εγώ να πω προς όλα τα μέλη της Επιτροπής ΔΕΒΕ, σας παρακαλώ βγείτε γρήγορα από την αίθουσα. So it was not on the micro we realized. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά καταλάβατε καλά.